Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Καταρχάς έχουμε κάποιες τροποποιήσεις στην ημέρησια διάταξη. Το σημείο 4. Αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής αναβάλλεται για μετά τις ψηφοφορίες στις 11.30. Σήμερα το πρωί πάντα. Και επειδή η συνδιαλλαγή που έγινε προχτές, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, τα μεσάνυχτα, δεν κατέληξα, η ψηφοφορία για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης και του Μέσου ε, Ευελιξίας, οι εκθέσεις Χριστοφόρου και Βιώτη αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση. Εφόσον βέβαια εντωμεταξύ θα έχει προκύψει συμφωνία για το σχέδιο προπολογισμού 2019. Ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης και τον κανονισμό σχετικά με το ΦΕΝΤΕΡ και το, το Ταμείο Συνοχής 14 και για τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις ε, σημείο 18 μου ρεσάν αναβάλλονται διότι έχει αναβληθεί ψηφοφορία στη Ρέτζη το 27 Ευρωπαϊκή συνοριαφυλακή και ακτοφυλακή θα συζητηθεί πριν το 26. NDE σε Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίθηκε η τροποποιηθήσα ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα εορτάσουμε την 70η επέτειο της ε, Παγκόσμια Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 από τα 58 κράτη-μέλη που ήταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν αύριο θα εορτάσει αυτήν την 70η επέτειο. Η επικαιρότητα μας υπενθυμίζει τακτικά αυτή την κληρονομιά. Οπότε οι δημοκρατικοί θεσμοί που είναι κληρονόμοι και θεματοφύλακες των ευρωπαϊκών αξιών και της ε, χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι λοιπόν δικό μας καθήκον να συνεχίσουν να ζουν και να ακτινοβολούν αυτές οι αξίες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα οργανώσει αυτή την τρέχουσα εβδομάδα την πρώτη εβδομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω λίγα λόγια όπως και οι πρόεδροι των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το θέμα αυτό. Φυσικά δεν έχει να κάνει με τις εργασίες τη Επιτροπής προπολογισμών να ασχοληθούμε άμεσα με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση. Ο προπολογισμό δεν είναι όμως ένα τυχαίο νομοθετικό έργο. Μέσω του προπολογισμού, κάθε κοινότητα εκφράζει και μετρά τις δυνατότητες να ε, επιτελέσει το στόχο της να πραγματοποιήσει το εγχείρημά της. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι κατά την ε, προετοιμασία των ετησίων προπολογισμών και του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή Προπολογισμών δεσμεύεται, ούτω ώστε ο ευρωπαϊκό προπολογισμό να εξυπηρετεί αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή δέσμευση για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ο προπολογισμό πρέπει να είναι η πιστή έκφραση των αξιών μας. Στα πλαίσια της Ένωσης, η Επιτροπή Προπολογισμών έχει περασπιστεί επαρκή χρηματοδότηση για τα προγράμματα ε, στον τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ηθαγένειας, για ε, ε, την ισότητα, την Ευρώπη για τους πολίτες και τις πρωτοβουλίες των πολιτών μας. Επίσης, το Κοινοβούλιο πάντα έχει επιμείνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της, ούτω ώστε τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των ατόμων κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού να γίνονται σεβαστά. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής συγκυρίας, το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλαμβάνει πάντα τις ευθύνες του και να συμβάλλει πλήρως για να αντιμετωπιστούν οι βίες πράξεις κατά των πιο ευαλότων στρωμάτων της κοινωνίας μας. Αν δεν έχουμε επαρκή παρουσία, αυτό θα ήταν ε, ομολογία ενοχής. Πρέπει λοιπόν ο προπολογισμό να ανταποκρίνεται στι φιλοδοξίε μα και να ικανοποιεί τι απαιτήσει των θυμάτων. Γι' αυτό πρέπει να επαρρυπνούμε ούτε ώστε ο προπολογισμό μα να είναι αρκετά τολμηρό. στο Κοινοβούλιο τόνισε ότι το επόμενο πολιετέ πλαίσιο θα πρέπει να προωθήσει ω θεμελιώδει αξίε την ειρήνη, τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φίλων. Γι' αυτό τον λόγο η Επιτροπή Προπολογισμών κινητοποιήθηκε και ζήτησε εκπεφρασμένα να υπάρξει ουσιώδης πολιτική για θέματα ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης. Να υπάρχουν επαρκή μέσα. Αυτά είναι ακριβώς στο πλαίσιο της ε, παγκόσμιας διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρώπη πρέπει να διαφυλάσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των συμπολιτών. Πρέπει να προστατεύουμε του συμπολίτε μα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τι βαθιέ αιτήσει τη μετανάστευση και των μετακινήσεων σε τρίτε χώρε και να διασφαλίσουμε επί τόπου το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, να προλαμβάνονται οι σειράξει και να υπάρχει προοπτική ανάπτυξη. Αγωνιστήκαμε ούτω ώστε οι διάφοροι οργανισμοί μα, τα προγράμματά μα και οι πολιτικέ τη Ένωση που συμβάλλουν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ε, καθώς και οι ε, έλεγχοι στα σύνορα να έχουν επαρκείς ε, δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη ροή προσφύγων. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που να αποδεικνύει την αλληλεγγύη της δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ειρήνη και την ευημερία στις χώρες προέλευσης, αποδίδοντας περισσότερη σημασία στις επενδύσεις και στις πολιτικές ανάπτυξης. Εκεί όπου υπάρχει ένδια, εκεί που υπάρχει ανυπομονησία, να παραμείνουν λοιπόν οι πληθυσμοί στις χώρες προέλευσής τους. Απαιτήσαμε και νομίζω ιδιαίτερα από την Τουρκία στα πλαίσια της ιδιαίτερης ε, διευκόλυνσης για την Τουρκία οι ευρωπαϊκοί πόροι να συνδυάζονται με βελτιώσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. 70 χρόνια μετά την έγκριση τη διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σαφέ ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μα και ότι σημαντική πρόοδος πρέπει ακόμη να επιτευχθεί με τις ε, δικές μας αρμοδιότητες η Επιτροπή μας έκανε ό,τι μπορούσε ούτως ώστε ο προπολογισμό της Ένωσης να συμβάλλει ένεργα ούτως ώστε να προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό λοιπόν οι πόροι για την έρευνα αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την πορεία μας αυτή και να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι θεμελιώδεις αρχές δεν θα είναι απλά λόγια, αλλά θα εφαρμόζονται συγκεκριμένα χάρη και μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών. Για να μπορέσει εκ νέου και η πολιτική και οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες μέσω των δημοσιονομικών πράξεων να αρθούν στο ύψος των διακηρύξεων τους. Σας ευχαριστώ πολύ. vous avez... λάβατε τα σχέδια πρακτικών των συνεδριάσεων τη 9η Οκτωβρίου και τη 5η Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι αυτά τα πρακτικά ενεκρίθησαν. Και τώρα να ψηφίσουμε σχέδιο νομοδότησης για το νομοθετικό πρόγραμμα του επομένου πολιετούς πλαισίου 21-27. Σας παρακαλώ ε, να κάνουμε έναν έλεγχο. Ε, βάλτε τις κάρτες σας στα μηχανήματα για να κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ε, λείπει μία ψήφος. Πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη ψηφοφορία. Έκθεση Αλή για το στρατηγικό ε, πρόγραμμα για την κοινή γεωργική πολιτική. 31 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 ε όχι Το 8 καταπίπτει λοιπόν ναι 34 που είναι συμβατή με το 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε άρχεται. Ελέγχουμε τη 10. Πέρας. Δεκτή. 19 υπέρ, 13 κατά και μία αποχή. 35 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτε 38 και 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 40 και 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 42-43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 44-45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 46, 47, 48 και 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται για την 11 Πέρασε. Δεκτή. 18 υπέρ, 16 κατά. 52 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Την 53. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά, 11 υπέρ. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12, 13, 14 και 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 έχει αποσύρθει. 59 υπέρ Είπα 59 τώρα. 59 είπα. Το 58 όντω έχει αποσυρθεί. Ή 58. Τώρα όμω είπα για την 59. Ψηφίζουμε την 59. Ε, κατά αποχέ απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλά, ελέγχουμε την 59. Ψηφίσατε όλοι μου. Πέρασε. Απορρίπτεται 12 υπέρ, 22 κατά. 60 ήρθε, 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 για τις συντολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 Α, κατά πίπτη 19, συγγνώμη. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 21 κατά πίπτη. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 22 τώρα. Με την προφορική τροπολόγηση. Υπέρ. Κατά Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26. Αποσύρθηκε. 27. Με την προφορική τροπολόγηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5 Α, ε, 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Το σύνολο του κειμένου τώρα όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίζατε όλοι. Πέρας. Δέκτη 27 υπέρτασης κατά και δύο αποχές. Συγχαίρουμε τον κύριο Αλή. Για την ε, έκθεση του συναδέλφου Κουσμιούτ σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική και τη διαχείριση και την παρακολούθηση. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 33 Ψήφισατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 15 κατά. 34 υπέρ. Qui contre, qui Απορρίπτεται 10 και 35 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 11 και τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. αποχές να επαληθεύσουμε για τις 11 και 5 τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 14 κατά. 36 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε γιατί 12. Ψήφισατε όλοι. <laughs> Υπάρχει μια κάρτα που έχει απομείνει μόνη τη. Λήξη. Απορρίπτεται. 18 κατά, 13 ψηφοί υπέρ. Ήταν η τροπολογία 12. Πάμε στην 13 και στην 6. Που έχουν το ίδιο αντικείμενο. Υπέρ. Κατά. Πιστεύω ότι απορρίπτεται για την 13 και την 6. Vote est clos. 17 voix Απορρίπτεται 17 κατά 15 υπέρ. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17, 18, 19 και 20 οι τροπολογίες αυτές υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 αποσύρεται. 24, 25, 26. ...24, 25, 26... Είπα και 27, αλλά όχι, 8 εννοούσα. 24, 25, 26 8. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 38, υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε για την 38. Λήξη. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 13 κατά. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Θέλετε επαλήθευση για την 28 άρχιτη ψηφοφορία. Για την 28 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται 17 υπέρ 15 κατά για τις αντιολογικές σκέψεις. Πάμε στην τροπολογία 29 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχουμε συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Έχουμε εδώ τμήματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Ποιος είναι υπέρ για την 32. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Έγκριση με 24 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 5 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε τώρα στην έκθεση Καρδία Σαμπάλ Περουμπιάλ. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Ελίας. Τροπολογία 42 και 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Να επαληθεύσουμε. Να επαληθεύσουμε τις 42 και 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Λήξη απορρίπτεται 17 κατά 13 υπέρ. Τροπολογία 13, 14 και 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 15 και 16 υπέρ. Και 17, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 43, 44, 45 και 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48, 49 και 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 50 και 51 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε για την 50 και 51 άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνονται. 17 υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 52 και 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Εποχέ, εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Εποχέ να επαληθεύσουμε για την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 15 κατά. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την 20. Λήξη. Απορρίπτεται 16 κατά 14 υπέρ. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές Συγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται 10. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 26. Καταπίπτει 26 γιατί εγκρίθηκε η 10. 27 υπέρ. Κατά αποχές Συγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 28 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε λήξη απορρίπτεται 18 κατά 12 υπέρ ήταν η τροπολογία 28 πάμε στην 29 υπέρ κατά αποχές Συγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Κοιτάξτε. Τώρα εδώ μόλις ψήφισαμε για την 33. Λήξη για την 33. Απορρίπτεται. 17 κατά 14 υπέρ. Θέλετε έλεγχο για την 31. Άρχεται ψηφοφορία για την 31. Λήξη. Απορρίπτεται. 19 κατά 12 υπέρ. 34 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη. Για την 34. Λήξη. Απορρίπτεται. 19 κατά 12 υπέρ. Περνάμε στην 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε Ήδη 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 17 έναντι 13. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται 40 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται 12 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται 41 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Για τις παραγράφους τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 3 άρχεται η ψηφοφορία λήξη απορρίπτεται 16 κατά 15 υπέρ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται 27 υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Καρδιζαβάλ. Τώρα θα ψηφίσουμε σχετικά με τη θέση του μηχανισμού προτεξιακής βοήθειας 3 Έκθεση Μάλετιτς. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 29 ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι, λήξη. Απορρίπτεται 19 κατά, 12 ψήφι υπέρ. Περνάμε στην 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 αποσύρεται, 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για τις αιτηλογικές σκέψεις 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε το 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται. 22.99, 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 20. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ συγγνώμη καταπίπτει 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για τα παραρτήματα Τριάντα τρία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές να παληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 35 λήξη απορρίπτεται 18 είναι το 13 36 υπέρ κατά απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Εγκρίνεται 27 υπέρ, Θα σας ψήφι κατά και δεν υπάρχουν αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Μάλετιτς. Τώρα, για την έκθεση τη δική μου, του Πρόεδρου. Εράσμους. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται, 22. Αποσύρεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Για τα εκτιμώντα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου όπως ε, τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται με 29 υπέρ, 2 κατά, δεν υπάρχουν αποχές ή χαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα έκθεση Τίμο Βέλκεν. για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά απόχέ, δεκτή. 9 και 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτές. Παραρτήματα 10 και 7 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Αιτιολογικές σκέψεις 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πέντε υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 με προφορική τροπολόγηση του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε ονομαστική άρχεται Πέρας. Δεκτή 27 υπέρ, 4 κατά και χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Τίμο Βόλκεν. Έκθεση δεύτερη μάλιστα του κυρίου Αλή, δεύτερη σήμερα το πρωί. Για το πρόγραμμα καταπολέμησης των απατών. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται άρχεται πέρας απορρίπτεται 14 ψηφί υπέρ 16 κατά. στο 8 ήμασταν. Α, ήμασταν στο 9. Α, στο 9. Θέλετε να ελέγξουμε και την 8. Καλά, να ελέγξουμε και την 8. Επαναρχόμεθα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 14 υπέρ, 17 κατά τροπολογία 1 υπέρ. Κατά εποχές, δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. δεν σαφές. Ελέγχουμε τη 2 παρακαλώ, άρχεται. Κοιτάξτε, δεν ε, σηκώνετε όλα τα χέρια οπότε ορίστε, τιμωρία. Πέρας. 28 υπέρ 3 κατά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ο απολογισμό ε, διοξείδιου του άνθρακα δεν είναι πολύ καλό. 10 ε, υπέρ κατά. Αποχέ. Δεκτή. 3 υπέρ κατά. Αποχέ δεκτή. Ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Άρχεται. Πέρας. 28 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Αλή. Λοιπόν, οι ψηφοφορίε θα συνεχιστούν σήμερα το απόγευμα, στις 3. Οπότε τώρα θα σας ενημερώσω για την ε, συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό. Η πρώτη της φάση ολοκληρώθηκε την ε, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό του 2019 θα πρέπει να επαναληφθούν ε, τις ε, αμέσως επόμενες μέρες αλλά, αλλά Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Γενικό Εισηγητή και τους εισηγητές για τα άλλα τμήματα και στον μόνιμο εισηγητή για τους εξωτερικούς οργανισμούς και να ευχαριστήσω και όλους και όλες όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις δυσάρεστες διαπραγματεύσεις όπου περνάει κανείς ατελείωτες ώρες περιμένοντας ε, τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ που μείνατε εκεί μέχρι το τέλος και παραμείναμε όλοι ενωμένοι στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο. Το οποίο Συμβούλιο τελικά απεδείχθη αδιάλακτο. Θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο Έτινγκερ για όλες τις προσπάθειες που έκανε για να επιτευχθεί ένα συμβασμός. Πρέπει να πω ότι μας εξέπληξε η κατάληξη γιατί είχαμε ξεκινήσει καλά. Σε ένα γεύμα την Παρασκευή 16 όπου ήταν μαζί μου ο κύριος Βιώτη, ο κύριος Ζούμπη και ο κύριος Γκάια. Είχαμε την εντύπωση ότι θα καταλήγαμε χωρίς ε, δυσκολίες πριν την λήξη του απογεύματος. Μετά όλα χειροτέρεψαν πολύ στα μέσα του απογεύματος για τη χρήση του νέου άρθρου 15.3 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού τον οποίο εγκρίναμε στις αρχές του τρέχοντος έτους και ο οποίος επιτρέπει οι πιστώσεις για την έρευνα όταν δεν έχουν δεσμευθεί πλήρως κατά το έτος N-2 ε, να χρησιμοποιηθούν για το έτος 1. Και ακούμε συνεχώς όλους να λένε ότι η έρευνα ε, είναι προϋπόθεση του μέλλοντός μας, η δυνατότητα να μην ε, είμαστε υποδέστεροι των γιγάντων της ψηφιακής οικονομίας της Κίνας και των ΗΠΑ να επανέλθουμε στην ψηφιακή μας κυριαρχία. Τότε όμω ε, αντιμετωπίσαμε μια ακαμψία από πλευρά Συμβουλίου. Ναι, μεν, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιχείρησαν να προσθέσουν νέο χρήμα για να καλυφθεί αυτή η έλλειψη 400 εκατομμυρίων που είχε να κάνει με την αναβολή ε, των, ε, της χρήσης του ορίζοντα για το 2017. Είναι εξτρέμις η Κομισιόν πρότεινε να μειωθούν οι περικοπέ σε άλλα προγράμματα, αλλά ήταν μόνο μερικέ δεκάδε εκατομμύρια που τα παίρνουν δεξιά-αριστερά. Δεν ήταν επαρκή. Και τίποτα δεν κινήθηκε για να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 15.3. Μόνο η πρόταση να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασία οπωσδήποτε υψηλού επίπεδου με εκπροσώπους του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου με επικεφαλή στον κύριο Μόντι ή από κάποιον ε, αυτού του επίπεδου. Κλασική αντιμετώπιση για να καταλήξουμε κάποτε σε μια απόφαση. Η Κομισιόν θα, θα υποβάλει συγγνώμη, νέο σχέδιο προπολογισμού που θα μπορούσε ίσως ε, να ε, φτάσει σε εμά ε, την Παρασκευή 30 τρέχοντος, δηλαδή σε 10 μέρες και η Κομισιόν στις 3 Δεκεμβρίου θα υποβάλει, θα παρουσιάσει την πρότασή της στις 2.30 στη συνεδρίασή μας και μετά θα έχουμε έναν ή περισσότερους τριμερείς ε, διαλόγους στις 3, 4, 5 ή και 6 Δεκεμβρίου. Και αν προκύψει τότε συμφωνία, το Κορεπέρ θα μπορούσε να το εγκρίνει στις 7 ε, και το Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου πάντα. Οπότε ο προπολογισμό του 19 θα μπορούσε να ψηφιστή στο Στρασβούργο. Και τώρα να δώσω το λόγο στο γενικό μας εισηγητή. Ντανιέλ Λεβιώτη ο οποίος επέδειξε απόλυτη συνέπεια στη θέση του, με βάση και την εντολή που είχε λάβει και από εμά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω τη ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί του σχεδίου προπολογισμού του 19 και με τη στήριξη τη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Ντανιέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως στην ε, συνεδρία της Ολομιλίας μας, στην ε, γραμματεία της Επιτροπής μας, στις πολιτικές ομάδες, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων που μας υποστήριξαν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά σε όλο το στάδιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού για μένα. Ήταν μια καινούρια εμπειρία προφανώς, μια πολύ σημαντική εμπειρία και σίγουρα θεμελιώδης, αλλά χωρίς την υποστήριξη όχι μόνο τεχνικού χαρακτήρα, αλλά και πολιτικού χαρακτήρα και ψυχολογική υποστήριξη, αν μου επιτρέπετε, της ε, γραμματείας ε, και του προσωπικού των πολιτικών ομάδων, θα ήταν πραγματικά δύσκολο να αντιμετωπίσω όλη αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και σας Πρόεδρε, αλλά και τους ε, συναδέλφους, συζητητές των υπόλοιπων τμήματων, αλλά και για τους οργανισμούς και του συναδέλφους που ήταν παρόντες και με υποστήριξαν πολιτικά καθόλου το στάδιο της συνδιαλλαγής. Δεν είναι δεδομένο να έχει κάποιος τόσο ισχυρή πολιτική στήριξη και υπενθυμίσατε εσείς ότι έπρεπε και να ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια των συνεδριασεών μας για να επιβεβαιωθεί η εντολή στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, προσπαθώ να πω στους συναδέλφους απλώς ποια είναι τα κύρια πολιτικά στοιχεία, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, που προκάλεσαν τις διαφορές και δεν μπορούσαμε να κλείσουμε την πρώτη συνδιαλλαγή είχαμε προβλήματα ε, επί της ουσίας και επί της αρχής. Τα προβλήματα επί της αρχής ε, στήσονται με δύο θεμελιώδη θέματα. Το ένα το συζητάμε από τον Ιούλιο και ε, το θέμα αυτό ακούγεται σε όλο το Κοινοβούλιο. Εμείς ποτέ δεν το αφαιρέσαμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το θέμα της χρηματοδότησης ε, για τον μηχανισμό ε, για τους πρόσφυγες στην ε, Τουρκία. Και μπορώ να πω, μέχρι τέλους σε κάθε επίσημη συνεδρίαση με τον Υπουργό, με το Συμβούλιο, και σε όλες τις ε, συναντήσεις ε, πάντοτε εμείς θεωρούσαμε ότι εξακολουθεί να παραμένει για μας αυτό το θέμα αρχής. Επίσης, ένα άλλο θέμα αρχής είχε να κάνει με την εφαρμογή του άρθρου 15.3 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Εμείς ζητήσαμε την εφαρμογή γιατί έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο, ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το δώσαμε στον εαυτό μας και μας επιτρέπει να λέμε δεν ζητάμε νέους σπόρους από τα κρατη αλλά χρησιμοποιούμε τους υφιστάμενους σπόρους, κυρίως για τα μέτρα που είναι τόσο σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης και για τα κράτη-μέλη, έρευνα και νέοι. Εμείς αυτό θέλουμε να αποκτήσουμε. Όμως το Συμβούλιο έδωσε μία απάντηση και η οποία ήταν εντελώς ε, κάθετη, ε, αλαζονική στάση. Δηλαδή προσπάθησε να επιβάλλει στο Κοινοβούλιο τις δικές του προτεραιότητες, να πούν σε εμά ποιες θα είναι οι δικές μας προτεραιότητες και να μας πούνε ποια είναι τα θέματα που μπορούμε να θίξουμε ή όχι. Και επανειλημμένα σε επίσημες συνεδριάσεις μας ζήτησαν να μην ανοίξουμε πλέον τη συζήτηση για το άρθρο 15.3 και για το μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, γιατί ε, τα κράτη-μέλη ε, θα τη δράσουν. Ε, κοιτάξτε, Πρόεδρε, εμείς ήμασταν όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί μπορούσαμε απέναντι στο Συμβούλιο στο στάδιο των συζητήσεων. Όσο πιο ανοιχτοί μπορούσαμε μάλιστα ακόμη και να συζητήσουμε θέματα που για μας ε, ε δεν ήταν συζήτηση, όπως πιθανές περικοπές, παραδείγματο χάρη μείωση ε, των αυξήσεων σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε μα. Όμω, εγώ ε, δεν ε, θέλω να μου επιβάλλουν ε, τη δική μου στρατηγική και να μου πούνε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Εμείς είμαστε συνομοθέτες στον προϋπολογισμό και έχουμε τα δικά μας επιχειρήματα και έχουμε το ίδιο κύριο στη συζήτηση με το Συμβούλιο για την συζήτηση. Και αν μου λέει το Συμβούλιο ότι είναι κάτι απαραίτητο και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τη δυσκολία για την εφαρμογή του 15.3 και για το μηχανισμό για την Τουρκία, εγώ δεν μπορώ να ε, αντιδράσω διαφορετικά παρά να πω ότι και για μας είναι εντελώς απαραίτητα αυτά τα θέματα, γιατί δύο τεχνικά θέματα γίνονται πολιτικά τελικά. Και να σας πω και δύο λόγια για το τι συμβαίνει τώρα, κατόπιν αιτήματος των συναδέλφων ε, της Επιτροπής. Θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους είναι προφανές ότι η συζήτηση η σημερινή δεν αφορά τον προϋπολογισμό του 2019, δεν αφορά μόνο τον προϋπολογισμό του 2019 η συζήτηση αφορά το συσχετισμό των δυνάμεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και συζητάτε το θέμα της ικανότητας να έχουμε εμείς ε, τα κατάλληλα εργαλεία και να τα δώσουμε στους συναδέλφους στο και Όλμπρεκτ στις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα έχουν για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η σοβαρότητα με την οποία εμείς θα προσεγγίσουμε το δεύτερο μέρος της συνδιαλλαγής και θα μείνουμε σταθεροί στις αρχές μας και στα αιτήματά μας επί της αρχής θα είναι τα εργαλεία και η αξιοπιστία με την οποία θα παρουσιαστούν στις διαπραγματεύσεις οι συνάδελφοι Τόμα και Όλμπρικτ και φυσικά και ο συνάδελφος Ντεπρέ και ο κύριος Λεβαντόφσκι για τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό διακυβεύεται. Δεν διακυβεύεται μόνο ο προπολογισμός του 2019. Ε, αυτό είναι το τελευταίο λοιπόν που λέω και η έκκληση που κάνω στην Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να συζητήσουμε εις βάθος για τη θέση μας, που θα πρέπει να είναι κάθετη και να εμείνει στις αρχές της κατά την άποψή μου στους συντονιστές αποφασίστηκε το άρθρο 15.3 να θεωρηθεί ως ένα κομβικό σημείο της συζήτηση με το Συμβούλιο. Εγώ έχω το προνόμιο να είμαι εισηγητής για τον προεπιλεξισμό του 2019 και έχω κάθε πρόθεση, Πρόεδρε, να κλείσω θετικά αυτό τον προϋπολογισμό, να τον κλείσω στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Εγώ θα εργαστώ όσε ώρε χρειάζεται και θα κάνω κάθε προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσω από του αδέλφους βουλευτέ να ψηφίσουν ένα προπολογισμό που αποκλίνει από τι αρχέ μα και δεν ανταποκρίνεται σε όσα ψηφίσαμε τον Οκτώβριο, στο Μάρτιο, στι κατευθυντήριε γραμμέ και στη θέση μα τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, κύριε Γενική Συγκητά. Ναι, ναι, μπορούμε και να τον χειροκροτήσουμε. Κοιτάξτε, πότε φαίνεται, εφαρμόζουμε στον τομέα της έρευνας το εξής. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς να το πω, να δίνουμε και να παίρνουμε. Λοιπόν, ας ακούσουμε και τον εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα. Αντικαθιστά ο Χωσημανώλη τον κύριο Ρούμπικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα κάνω και άλλα σχόλια, όχι μόνο για το τμήμα 5, που αφορά τον κύριο Ρούμπιχ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές, το Γενικό Εισηγητή, αλλά και τον εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει την ενότητά του και είναι ένα θέμα δικαιοσύνης αυτό που υπερασπίζουμε. Επίσης, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, ελπίζω, ότι ο Επίτροπος δεν θα υπαναχωρήσει τώρα μπροστά στην αδιαλαξία και στην παράλογη θέση του Συμβουλίου. Να υπενθυμίσω, πρόκειται για ένα προπολογισμό 0,9% του εθνικού ακαθαρίστου εισοδήματο και δεν σέβεται το Συμβουλίο τις συνθήκες δεν αναγνωρίζει τον κανονισμό που υιοθετεί. Το Συμβούλιο είπε με λεζονία ότι το Ταμείο για τους πρόσφυγες την Τουρκία είναι 2 δισεκατομμύρια για τον προπολογισμό και ένα δισεκατομμύριο για μας και αυτό δεν αλλάζει. Είναι κάτι αμετάκλητο. Πήρε τις αρμοδιότητες στην εξουσία του Κοινοβουλίου και επίτηδες ξέχασε ότι και εμείς ε, είμαστε ε, δημοσιονομική αρχή. Λέει το Συμβούλιο, ο προπολογισμό είμαστε εμείς. Στη συνέχεια υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη που θέλουν να πούν όχι εγώ είμαι ο προπολογισμό. Αυτό που κάνουν ε, κάποια, αυτό κάνουν κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με τη θέση τους σχετικά με την έρευνα. Εμείς Υιοθετήσαμε έναν δημοσιονομικό κανονισμό και πραγματικά εκπλήσωμε. Το Συμβούλιο δεν έχει καταλάβει τι έχει υιοθετήσει. Το Συμβούλιο τώρα αμφισβητεί τον ίδιο τον κανονισμό που υιοθέτησε. Λοιπόν, ε, το να μιλάμε για το 15.3 δεν σημαίνει τίποτα. Οι πολίτες ε, όμως κατανοούν ότι το Συμβούλιο θέλει να πετάξει εκτός 413 εκατομμύρια που είχαμε για την έρευνα. Αυτά τα 413 εκατομμύρια είχαν δεσμευτεί αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Το κοινοβούλιο θέλει κάτι πολύ απλό. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την έρευνα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για την Ευρώπη, για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση. Και υπάρχει κάτι ακόμα που πιστεύω ότι δεν ξέρουν οι πολίτες. Ο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την έρευνα όταν η Γερμανία είναι η χώρα που χρησιμοποιεί περισσότερο την έρευνα. Οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες ξέρουν ότι ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας τους δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τους πόρους για την έρευνα και μιλάμε για πόρους διαθέσιμους. Οι Γάλλοι πολίτες ξέρουν ότι ο Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που για την έρευνα. Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα που χρησιμοποιεί περισσότερο τα κονδύλια από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και δεν είμαι και σίγουρος αν ο Εμμανουέλ Μακρόν ξέρει ότι είχε έναν υπουργό που παρά τις προτάσεις που κάνει για περισσότερη Ευρώπη τελικά θα αυτές τις θέσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά. Το Κοινοβούλιο δεν έχει ζητήσει τίποτα ιδιαίτερο. Το Κοινοβούλιο έκανε τα πάντα για την επίτευξη συμφωνίας. Και υπάρχει κάτι που με ανησυχεί. Με την αλαζονία του Συμβουλίου με τη θέση ότι ο προπολογισμό είμαστε εμεί, με τη θέση κάποιων κρατών μελών. Όχι, ο προπολογισμό είμαι εγώ. Το Συμβούλιο προσπαθεί ε, ουσιαστικά ε, να μπορεί να εκμεταλλευτεί το ίδιο το 1 12 Και τι γίνεται με το Brexit, δεν αρκεί το πρόβλημα του Brexit. Θέλουν να προσθέσουν προβλήματα το Συμβούλιο θέλει να δώσει επιχειρήματα στους λαϊκιστές, τους εξτρεμιστές, τους ακραίους, για να λένε ότι τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Και γιατί μιλάμε για τίποτα, για 0,01 του προπολογισμού ή ούτε καν. Και το Συμβούλιο με τη στάση αυτή κάνει ένα δώρο στους εξτρεμιστές για να πούνε σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και τώρα και άλλα επιχειρήματα για να αμφισβητήσουμε την Ευρώπη και το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι θρελό και να ζητήσει η αλλαγή των συνθηκών για να πει ότι το Συμβούλιο μόνο καταρτίζει το προπολογισμό και το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία φωνή για το θέμα αυτό. Αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε και να δείξουμε στους πολίτες ότι θέλουμε ένα προϋπολογισμό και ότι το Συμβούλιο κάνει τα πάντα για να μην υπάρξει προπολογισμό. Και θα πω και κάτι ακόμη. Δεν ε, θα εκπλαγώ αν τελευταία στιγμή έρθει το Συμβούλιο με άλλες προτάσεις λαϊκιστικές για να πει το κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη, δεν ήθελε να κάνουμε εξοικονομήσει, ε, παραδείγματο χάρη για τον τομέα 5 κτλ πάντοτε προσπαθεί να αποφύγει την επίτευξη συμφωνίας. Και σίγουρα αυτή η θέση δηλώνει ασέβεια απέναντι στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν σέβεται ούτε στους πολίτες, ούτε τις διακηρύξεις του ίδιου του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στους Κιώδης τώρα. Ο Χωσέ Μανουέλ ε, ε, εκπροσωπούσε την κυρία Χόλμαια. Ο κύριος Χόλμαια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το διεξοδικό τους έργο και την επιμονή την οποία επιδεικνύουν. Φετέρου βεβαίως γνωρίζετε ότι η πολιτική ομάδα ECR ε, έχει άλλες πολιτικές θέσεις. Γνωστές είναι, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Γι' αυτό και θα ε, αρκεστώ σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόλμελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που τόσο θαυμάσια παρουσίασε ο συνάδελφος ε, Ζωζέ Φερνάντες. Και δεν είναι κάτι έτσι τυπικό, κάτι που βαθιά πιστεύω. Η αντιπροσωπή του Κοινοβουλίου με τον κύριο Βιώτη με εσά ε, ε, κατέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μια απόλυτη ενότητα που είναι ουσιώδες στοιχείο. Η θέση του Κοινοβουλίου όντως ήταν η βάση των προσπαθειών μας. Ο Ζωζέ Μανουέλ είπε ότι ε, ορισμένοι θεωρούν και ίσως να το πιστεύει ο κ. Κόλμερ ότι αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να υπάρχουν υπερβολικέ δαπάνε. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Εμεί θέλουμε μόνο 1% στι ε, δεσμεύσει και 0,9% στις ε, πληρωμές του ακαθάριστου του εθνικού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν πολλά προηγούμενα στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο προπολογισμό είναι τόσο λίγο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο. Άρα δεν μπορεί κανεί να πει ότι είμαστε σπάταλοι. Και όπως είπε και ο Ντανιέλε, η επίσημη ε, πολιτική ε, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, συγγνώμη, το καθιστά σαφές ότι δεν δέχονται το 15 τώρα γιατί δεν ε, θεωρεί, θεωρούν ότι η συζήτηση αφορά μόνο το προβλήμα του 19, αλλά και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλω να μα κλείσουν την πόρτα όχι μόνο για το 19, αλλά και κάτι πολύ ουσιώδε που οι συγκητέ μα το έχουν τονίσει. Δηλαδή να υπάρξει ένα αποθυματικό που να δημιουργείται από τι αποδεσμεύσει. Η δική μου ανάλυση τη κατάσταση στην οποία είμαστε τώρα είναι η εξή. Το αρνούνται αυτό γιατί θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το πολιτέ πλαίσιο. Στην οποία διαπραγμάτευση το Συμβούλιο θα εμείνει επί ιδιαίτερα αδιάλακτων θέσεων όσον αφορά τα ποσά. Η Επιτροπή προτείνει 1,08 εμείς απαιτούμε 1,3 δεν θα μας το δώσουν δεν θα μας δώσουν ούτε το ένα ούτε το άλλο η μόνη δυνατότητα να δημιουργηθούν ε, τέτοιες δίκες που να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις είναι να έχουμε και ένα μέγιστο ευελιξίας και αποθεμάτων και αποθεματικού και ιδίων πόρων. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι η στρατηγική μας. Γι' αυτό, κάτε Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι η Επιτροπή μας σήμερα πρέπει να δώσει εντολή και σε εσά και στο Γενικό Εισηγητή μα για να στείλουν ένα σαφέ μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα επιφορτιστεί με τη νέα πρόταση. καλώντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει ότι ούτως ή άλλως η ιδέα για τη χρήση του 15-3 ήταν δική της θέση. Δεν ήταν δική μας πρόταση, ήταν δική της. Εμείς βεβαίως την υιοθετήσαμε αμέσως, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα ευφύης πρόταση και ήμασταν ευγνώμονες. Δεν θα μας ζητήσετε τώρα να την εγκαταλείψουμε, αυτό θα τους πούμε. Και γιατί θεωρούμε ότι είναι καλή πρόταση, αλλά και γιατί ξέρουμε στα πλαίσια ποιας λογικής εγγράφεται. Οπότε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσουμε εντολή και στον Πρόεδρο και στον Γενικό Εισηγητή να πούν στην Κομισιόν ότι μια πρόταση που δεν θα περιλαμβάνει το 1053 δεν θα κριθεί από εμά. Ευχαριστώ κύριε Ντούπρε. Μα ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Γενικό Διευθυντή Κόπμαν είναι παρόν και θα δώσουμε το λόγο συντόμω. Η κυρία Νίρη Άντα δεν είναι εδώ. Ο κύριο Σολέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές και τον πρόεδρο της Επιτροπής μας που επέμειναν μέχρι τέλους και υπερασπίστηκαν την εντολή που τους δώσαμε ομόφωνα ως αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι εμείναμε στις θέσεις μας και ήταν ε, αναγκαίο να γίνει αυτό. Γιατί μπορεί να φαίνεται γελίο να μαλώνουμε για μερικές εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ευρώ σε έναν ε, ε, προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα δεν μιλούσαμε για αυτά τα εκατοντάδες Στι λίγε εκατοντάδες εκατομμύρια. Το αντικείμενο της συζήτηση ήταν ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη στον προπολογισμό και ε, την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων όπως έχουν θεσπιστεί. Και εδώ μιλώ για το δημοσιονομικό κανονισμό. Και το άρθρο 15 παράγραφος 3. Το άρθρο αυτό ισχύει, είναι εφαρμοστέο και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τεχνικά εμπόδια τόσο μεγάλα ώστε να μην μπορούν να ξεπεραστούν. Ώστε να χρησιμοποιείται αυτό ως δικαιολογία για να μην εφαρμόζεται ο κανόνας αυτός, η διάταξη αυτή. Επίσης πιστεύω ότι σε επερχόμενες διαπραγματεύσεις ε, για το πι-δελτα-πι ε, θα αντιμετωπίσουμε παρόμοια θέματα γιατί όλοι έχουν λάβει τις θέσεις τους για την επόμενη μάχη και ορθώς και δικαίως αλλά αυτό σημαίνει ότι και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να εμείνουμε στην ε, θέση μας για τον προϋπολογισμό του 2019 αλλά και για ό,τι πρόκειται να έρθει αργότερα. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Ντεπρέ και την έκκλησή του να αποστείλουμε σαφές μήνυμα στην Κομισιόν ότι στο επόμενο σχέδιο προπολογισμού θέλουμε πρόταση για το 15-3 Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση αυτή και θα υποστηρίξουμε και εμείς από την πλευρά μας την πρόταση αυτή. Ε, ευχαριστώ κύριε Σολέ. Σολτέκ. Α, αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε τότε η κυρία Καρθιαδάβαλ, η συνάδελφοι τώρα που είχα ζητήσει το λόγο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί πολλοί συνάδελφοι είπαν ε, αυτά που ήθελαν να πω. Γιατί όλοι συμφωνούμε. Μετά από δύο προσπάθειες, την Παρασκευή και την Δευτέρα, απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις. Καλά, όλοι είπαμε ότι δεν είναι δραματικό, ότι υπήρχε χρόνος, ότι θα υπάρξει νέα πρόταση Έχουμε μέχρι την 31η ε, Δεκεμβρίου για να συζητήσουμε μια νέα πρόταση. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι εγώ ανησυχώ. Γιατί όπως υπόθηκε συζητάμε για ένα προϋπολογισμό που είναι στο 1% του ακαθάριστου εθνικού ε, εισοδήματος. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα φιδωλοί. Και τι διαπιστώνω το Συμβούλιο είναι ε, αχόρταγο. Αν ήταν στο 1,1 θα ήθελε το 1. Ήμασταν στο 1 θα ήθελε το 0,9. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις πιστώσεις για κάποια προγράμματα να κάνουμε αλλού περικοπές. Αν χάσουμε χρήματα γιατί δεν ε, ε, χρησιμοποιήθηκαν πάνε χαμένα. Πρόκειται για μια περιδίνηση ε, απόλυτα παραλόγων περικοπών. Στην ουσία αυτό που δίνουμε είναι επιχειρήματα στους ε, λαϊκιστές. Εμείς στην ουσία απογοητεύουμε όμως και τους φίλους της Ευρώπης. Γιατί αυτό που απαιτούν δεν το βλέπουν. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Πολύ περισσότερο. Και ανησυχώ γιατί όπως λέγαμε και την Παρασκευή ίσως την Παρασκευή να είμαστε ανυπεραισιόδοξοι αλλά έχουμε πολύ ευνοϊκές ε, προϋποθέσεις, ε, κάτι που δεν υπήρχε το 18 ή τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πολύ περισσότερες δυσχέρειες που δυσχέρναν τη διαπραγμάτευση. Είχαμε πολύ σαφές προτεραιότητες και είχαμε πει ότι το Συμβούλιο έχει μια σαφή προτεραιότητα που είναι η τα προηγουμενα χρονια ειχαμε πολυ περισσοτερες δυσχερειες που δυσχερναν διαπραγματευση ειχαμε πολυ σαφες προτεραιοτητες και ειχαμε πει οτι το συμβουλιο εχει μια σαφη προτεραιοτητα που ειναι η διευκολυνση για την Τουρκία, εμείς έχουμε τις δικές μας, ε, θα μπορέσουμε κάπου να συμβιβαστούμε, κάπου που να γίνονται σεβαστές οι προτεραιότητες και των δύο πλευρών. Και επιπλέον σεβόμενοι το επίπεδο δαπανών που προέβλεπε το σχέδιο της Επιτροπής. Και όλα αυτά γιατί ακριβώς μας είχε δώσει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτές τις 400, αυτά τα 400 τόσα εκατομμύρια που μας επέτρεπαν να αυξήσουμε τις δαπάνες για την έρευνα και τον ορίζοντα 2020 που ήταν οι προτεραιότητές μας επαναχρησιμοποιώντα χρήματα που αλλιώ θα πήγαινε χαμένο. Χαμένα. Είχαμε λοιπόν όλα τα στοιχεία για να καταλήξουμε ε, σύντομα σε μια λογική συμφωνία. Και επειδή το Συμβούλιο είναι αχόρταγο, δεν θέλει να προχωρήσει τίποτα. Είναι τόσο τσιγκούνικο. Κόβει από εδώ, κόβει από εκεί. Δεν θέλει να αξιοποιήσει ε, δυνατότητες που μας δίνει ο δημοσιονομικός προϋπολογισμός που μόλις εγκρίναμε και που υπήρχαν στην ε, κοινή διακήρυξη. Επί ένα χρόνο τον ε, συζητούσαμε αυτόν τον προπολογισμό. Και τώρα θα κάνουμε μια επιτροπή, ε, μια ομάδα εργασία για να δούμε πώ θα εφαρμοστεί. Μα αυτά είναι ντροπή. Αν δεν θέλει να εφαρμόσει το δημοσιονομικό κανονισμό το Συμβούλιο, α το πει. Είναι δικαιωμάτων. Μια πολιτική απόφαση. Αλλά να πούν σαφώ ότι είναι διατεθειμένοι να πάνε χαμένα 400 εκατομμύρια για την έρευνα. Για πολιτικού λόγου. Να μην έρχονται τώρα μετά να μα λένε με νομικήστικα και τεχνικήστικα επιχειρήματα ότι θα πάνε χαμένα. Α το κάνει. Αν θέλουν να το κάνουν εμεί δεν συμφωνούμε. Εμεί από την αρχή τη ε, διαπραγματεύση του πολιετού πλαισίου είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλε τι δυνατότητε και αυτή είναι πολιτική δέσμευση και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα χρησιμοποιήσουμε όλε τι δυνατότητε, όλα τα εργαλεία ούτω ώστε σε ένα πολύ περιορισμένο πολιτέ πλαίσιο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ κατά την εκτέλεση. Και έχουμε ένα δημοσιονομικό οργανισμό που μα το επιτρέπει μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε αυτά τα 300 εκατομμύρια. Αν δεν το θέλει το Συμβούλιο, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Αλλά εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι να λέγω τέτοια πράγματα. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τι προτεραιότητέ του. Έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε και για λόγου διατήρηση των αρμοδιοτήτων μα ω αρχή επί του προπολογισμού, αλλά και για λόγου ε, πολιτική νομιμοποίηση. Και ελπίζω η Κομισιόν να μα ακούει προσεκτικά να λάβει λοιπόν υπόψη τις προτεραιότητε και των δύο οργάνων. Ο καθένα έχει τη δική του λογική, τη δική του εσωτερική λογική, τις δικές του πολιτικές προτεραιότητες. Όλα αυτά είναι απόλυτα συνδυάσιμα. Μια πρόταση, για παράδειγμα, όπως ε, μας κάνανε προηγουμένω. στη δεύτερη εκδοχή. Ήταν μια πρόταση που με μικρέ προσαρμογέ συνέπεπτε απόλυτα με την πολιτική βούληση των δύο οργάνων. Ευχαριστούμε για αυτές τις κάθετες σταθερές παρατηρήσεις. Ο κύριος Αντιπρόεδρος Σαβάρμα έχει το λόγο. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν. Ξέρω ότι τώρα είναι ε, η ώρα να υψώσουμε τη φωνή μας και να ξεκαθαρίσουμε στους, ε, στα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να προσφύγουμε και εναντίον του Συμβουλίου για το γεγονός ότι δεν θέλει να τηρήσει ε, κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να το πω ξεκάθαρα. Έχω την αίσθηση ότι η Κομισιόν μπορεί να προτείνει κάτι το οποίο θα δηλώνει ξεκάθαρα με δεσμευτικό τρόπο ότι το 15.3 του δημοσιονομικού κανονισμού θα εφαρμοστεί εν ευθέτω χρόνο. Αν αυτό συμβεί, σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αλλά προτού αυτό καταγραφεί επίσημα, εγώ λέω να υψώσουμε τη φωνή μας και να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα επηρεαστούν το Εράσμους, ορίζοντας 2020. Εμείς φυσικά δεν έχουμε καμιά τέτοια πρόθεση, αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε ε, κόκκινες γραμμές. Ακόμη και αν κατηγορηθούμε ε, στη συνέχεια. Αν δεν λάβουμε αυτή την ξεκάθαρη διατύπωση για το 15 που θα εφαρμοστεί το 2020. Γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο θέμα για εμάς. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ κύριε Σαβάρμα. Ο κύριος ε, Γκάιερ ήρθε. Έπρεπε να πάρει το λόγο για τους εξωτερικούς οργανισμούς. Ε, να δώσω το λόγο λοιπόν στο μόνιμο εισηγητή για τους εξωτερικούς οργανισμούς. Που θα μας ε, αναφέρει τα κονδύλια που αφορούν τους οργανισμούς. Ναι, με συγχωρείτε. Είχα ένα πολύ σημαντικό εξωτερικό ραντεβού. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, ε, είμαι κάπως διχασμένος, διότι την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία, σε λύση. Και μετά για προσωπικούς λόγους δυστυχώς ε, χρειάστηκε να εγκαταλείψω τις διαπραγματεύσεις. Είδα εν τέλει τα έγγραφα της Δευτέρας όπου υπάρχουν ε, ε, έγγραφα της Κομισιόν η οποία, τα οποία αποδεικνύουν ότι τελικά ξαναξεκίνησε η συζήτηση για τους οργανισμούς που εγώ νόμιζα ότι είχαμε καταλήξει σε συμφωνία. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχαμε συμφωνήσει στην ομόφωνα τη μείωση των, ε, της χρηματοδότησης για την ΕΑΖΟ κατά 9 ε, εκατομμύρια. Στο, στην τελική πρόταση της Κομισιόν στα έγγραφά της τελικά εμφανίζονται μείωση 69 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, είχα την, είχα την αίσθηση ότι είχαμε καταλήξει εκεί όπου υπάρχει συμφωνία, σε αυτό το πολύ μικρό τμήμα του προϋπολογισμού, θεωρούσα ότι δεν θα ξαναετίθετο ε, σε υποαμφισβήτηση αυτό. Αλλά αφού το ξαναθέτει η ίδια η Κομισιόν, ε, είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, και να το ξαναδούμε το θέμα όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα των όσων προβλέπει. Εγώ ανοιχτός είμαι και πρόθυμος να τα ξαναδώ και να δούμε και διάφορες δαπάνες και υπό το φως της, του επίγοντος ε, χαρακτήρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται όλα τα χρήματα να είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα Ιανουαρίου κατευθείαν, αλλά ε, το να επιτεθεί ο προπολογισμό ή τέλο πάντων να περικοπεί ο προπολογισμό τόσο δραστικά ενό οργανισμού, ε, αυτό δημιουργεί πραγματικά ε, προβλήματα. Και εδώ ε, αυτό αυτά θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Κατά τα άλλα, ε, νομίζω ότι ήταν κοινή η στάση γύρω από τους υπόλοιπους οργανισμούς μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, αν και η θέση του Συμβουλίου ήταν πάντοτε ότι όλα αυτά που συζητούμε δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, οριστικά. Ε, αλλά ότι ε, πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες ε, έχουν καλές πιθανότητες εφαρμογής. εφαρμογής. Τώρα, αφού τα πάντα έχουν μηδενιστεί και αφού περιμένουμε καινούριο σχέδιο προϋπολογισμού, προφανώς και όλα όσα είχαν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής ακυρώνονται. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Αυτό βέβαια τώρα είναι καθήκον των, των αξιωματούχων της Κομισιόν ε, αν θέλουν δηλαδή να ξαναδούν πράγματα ε, ε, για τα οποία είχαμε συμφωνήσει ή αν θέλουν να αλλάξουν και αριθμητικά στοιχεία. Βλέπω ότι γνέφεται καταφατικά, οπότε φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και να κλείσουμε με τους Κιώδης. Η Μόνικα πήρε το λόγο πριν, αλλά μπορεί να συμπληρώσει το σχόλιο του Ζωζέ και ο κύριος Τάραντ επίσης είναι σκιώδης. Η κυρία Τόμα, θα πάρει το λόγο μετά τον κύριο Τάραντ. Εγώ πήρα το λόγο στις, στους συντονιστές μόνο. Απλώς θέλω να προσθέσω το εξής. Πρώτο σημείο που δεν το έχουμε θέσει στο επίκεντρο της προσοχής μας επαρκώς είναι ότι το Συμβούλιο έχει πρόθεση να κάνει μαζικές ε, περικοπές στο τμήμα 5. Πάνω από 50 εκατομμύρια δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, διότι ε, αν περικόψεις τόσο πολύ τη διοίκηση, ώστε να μην μπορεί μετά η διοίκηση να τα εφαρμόζει, ε, τότε γιατί θεσπίζουμε νομικές πράξεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Χρειάζεται ε, ένας οργανισμός, μια διοίκηση να είναι στελεχωμένη για να μπορεί να αναποκρίνεται στα καθήκοντά της. Αυτό λοιπόν φαντάζομαι ότι θα ληφθεί υπόψη και στο νέο σχέδιο προπολογισμού που θα υποβάλει η Κομισιόν, ε, και θα ε, αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις που ασκούν οι λαϊκιστές. Το 2014 εγώ συμμετείχα σε, στον προπολογισμό που επίσης είχε ε, αποτύχει, όπου είχαμε αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις ως Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε και Τανιέλε και οι άλλοι συντονιστές και οι σκιώδεις θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε αν η Κομισιόν υποβάλει πρόταση χωρίς 15-3 τι φανταζόμαστε ότι θα κάνουμε. Ε, γιατί εγώ αυτή την αίσθηση έχω τι θα κάνει η Κομισιόν, τι θα κάνει το Κοινοβούλιο αν ε, προκύψει μια τέτοια κατάσταση. Θυμάμαι ότι το 2014, όπου η κυρία Γεωργίευα ε, ήταν τόσο ε, επιθετική και επίμονη που εμείς ίσα που καταφέραμε να κρατήσουμε τα, τα μπόσικα. Αλλά νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ε, για κάθε ενδεχόμενο γιατί η αλλαγή στάσης, η μεταστροφή ήταν, ήταν πολύ εμφανής το, την Παρασκευή. Πρώτα το, το, το Κοινοβούλιο λοιπόν καλείται να υπερασπιστεί και στη συνέχεια κατηγορείται για το γεγονός ότι υπερασπίστηκε τις αρχές του τις οποίες είχε, στις οποίες είχε καταλήξει. Το, το ζήσαμε το 2014, δεν έχω καμία όρεξη να το ξαναδούμε και τώρα. Το να μας παρουσιάσουν δηλαδή στη συνέχεια οι συνομιλητές μας ως μαξιμαλιστές. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια σαφή διατύπωση για το 15-3. Αν αρνηθεί η Κομισιόν, τα πράγματα ε, δεν θα είναι εύκολα, θα πρέπει να, να επιμείνουμε, αλλά θα πρέπει να, να, έχουμε και ε, αυτό στο, ε, στο, στο νου μας, στο μυαλό μας. Έχω την αίσθηση ότι η η Κομισιόν δεν θα υποβάλει πρόταση το 15 Ε, νομίζω ότι ε, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με την κυρία Γεωργίευα. Ξαφνικά είχε ξεχάσει στο δεύτερο γύρο ε, διαπραγματεύσεων αυτό που ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη στην πρώτη. Δεύτερον, για την πρόταση της Κομισιόν νομίζω ότι υπήρχαν 46 εκατομμύρια και αν εφαρμοστεί το, το Δουβλίνο 3 να ρυθμιστούν τα ζητήματα μέσω διορθωτικού, ε, διορθωτικού προπολογισμού. Ε, ο Έτιγκερ ε, το δήλωσε ξεκάθαρε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να έρθει εντός του 2019. Δεν το ανέφερε όμως αυτό το θέμα καθόλου στην τελευταία, στον τελευταίο γύρο διαπραγμάτευσης ότι θέλει να κάνει μια, μια πλήρη απαλυφή. Ε, είχαμε τη διαβεβαίωση ότι το Δουβλίνο 3 δεν πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή εντό του 19. Το λέω αυτό ενημερωτικά, αλλά σου το λέω ε, διότι η, η Κομισιόν θα πρέπει να, να έχει και αυτό ως στοιχείο, ως ένα το κρατούμενο αν θέλετε, ε, στο νέο σχέδιο που θα υποβάλει, να μην ξαναρχίζουμε από την αρχή. Ε, και αυτό ενδεχομένως θα ήταν καλό να επισημανθεί και να υπενθυμιστεί στον κύριο Έτινγκ. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Τάραντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Βασικά, εγώ είχα να πω παρόμοια με αυτά που είπε ο κύριος Σολέ, τον υποστηρίζω και θέλω να δώσω και το χρόνο αγορευσής μου στην ε, κυρία Τομά που σίγουρα έχει πολλά να πει. Μάλιστα καθώς σας έχουμε μεταβιβάσει το λόγο ήδη κυρία Τωμά. Απλώς να σας ευλογήσω, κυρία Τωμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Ταράν. Να πω ότι συμφωνώ και υποστηρίζω τα όσα υπόθηκαν για την ενότητα της αντιπροσωπείας, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι και για τη συνοχή της θέσης μας. Και Εγώ ε, μιλώ για τον πρόεδρο και για τους εισηγητές. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι περήφανο για την αντιπροσωπεία του και για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία, κατά την απόψή μου. Το πρώτο, όπως είπε και ο κ. Δεπρέ, αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι το ανέφερε και ο κ. Βιώτη αυτό. Εδώ έχουμε έναν συσχετισμό δυνάμεων που ε, ίσως να σκίσει κάποια πίεση στη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2019, όμως ε, προσοχή, δεν είναι πρώτη φορά διάλεκτο το Συμβούλιο. Όμως ε, το επιχείρημα που είναι ιδιαίτερα σαφές και το είδαμε και στην ανακοίνωση του Συμβουλίου αφορά το απόθεμα για την αποδέσμευση πιστώσεων και ίσως ε, μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή του 15.3. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, εδώ και καιρό δεν είναι νέο στοιχείο στη συζήτηση μεταξύ της Κομπισιόν και του Κοινοβουλίου αφενός και του Συμβουλίου αφετέρου. Και στην ανακοίνωση του Συμβουλίου λέγεται σαφέ, σαφώς, ωστόσο το Συμβούλιο ανησυχεί ότι αυτό θα δημιουργήσει προηγούμενο και υπάρχει αβεβαιότητα για τις συνέπειες για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν αυτή την γραπτή φράση, είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει να απαντήσουμε. Όμως αυτό υπόθηκε και πριν. Εγώ υποστηρίζω τα όσα είπε ο κύριος Ντεπρέ, να σταλεί μια επιστολή στην Κομισιόν που να λέει ακριβώς ότι με ικανοποίηση αντιμετωπίζουμε την πρόταση της Κομισιόν που μας ε, βγάζει από το διέξοδο και δεν θέλουμε επαναχώρηση όταν ε, μιλάμε για την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και του προϋπολογισμού. Αυτό είναι το πρώτο. Εγώ Υποστηρίζω την πρόταση του Ζεράρ Ντεπρέ να στείλουμε αυτή την επιστολή στην Κομισιόν για να πούμε ότι την υποστηρίζουμε και το λέω για το 19 αυτό το προσθέτω, όχι για το 2020. Γιατί πάντοτε αναβάλουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Όμως στην πραγματικότητα <laughs> οι υποσχέσεις αυτές απλώς δεσμεύουν αυτούς που τις ακούνε. Δηλαδή, ουσιαστικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι υποσχέσει για το 2020, κοιτάξτε, Εμεί μπορεί και να μην είμαστε εδώ και μπορεί να μα ενδιαφέρουν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμοστούν το 2019. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο, Πρόεδρο, θέλω να επιμείνω στην ε, ανακοίνωση του Κοινοβουλίου. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, θα βιαστώ, θα τα πω γρήγορα είχε υποθεί από το Συμβουλίο όλοι να είναι λογικοί στις ανακοινώσεις του και να μην επιτίθενται στο άλλο θεσμικό όργανο. Το Κοινοβούλιο απολύτως έχει σεβαστεί αυτή τη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και θα σας διαβάσω τον ανακοινώθεν τύπου που ακολουθεί αυτή τη γραμμή απολύτως. Ο καθένας έχει κάνει αξιέπαινες προσπάθειες ε, για τη συνδιαλλαγή κτλ. Πολύ ωραία εμείς σεβαστήκαμε Τώρα, το Συμβούλιο τι λέει στον κοινό τύπου. Ωστόσο, το Συμβούλιο έκανε μια επικοδομητική προσφορά κτλ. Και το Κοινοβούλιο προτίμησε να χρησιμοποιήσει κτλ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Εμείς ε, σεβόμαστε τις δεσμεύσει μα ενώ το Συμβούλιο όχι. Τι προτείνω λοιπόν. Να μην γίνουμε περισσότερο επιθετικοί, αλλά να είμαστε πιο διαφανείς. Εγώ θα ήθελα καθώς ε, δέχεται επίθεση στο Κοινοβούλιο στον κοινοθεντή που να πούμε στο Συμβούλιο, ακούστε, δεν είναι εδώ θέμα ποιο θα επιτεθεί σε ποιον, αλλά πρόκειται περί θέσεων που δεν φαίνεται ότι μπορούν να συμφιλωθούν αυτή τη στιγμή και να ποιε είναι οι θέσει μα με απόλυτη διαφάνεια. Νομίζω ότι θα κατορθώναμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση όπου φαίνεται το Συμβούλιο να παίζει τον καλομαθητή ενώ δεν είναι έτσι. Μάλιστα, θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ο κ. Κοπάνο εδώ παρόν από την αρχή της συνεδρίασης και είμαι σίγουρος ότι έχει καταγράψει τη θέση μας. Απλώς να πω ότι τα 12 το Συμβούλιο από την πλευρά του θέλει ένα δις για το μηχανισμό για την Τουρκία. Όταν ε, δεν υπάρχει προπολογισμό, δεν υπάρχει δισεκατομμύριο για την Τουρκία και πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και αν ε, θέλουμε ε, να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει και αλληλοσεβασμός. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, υπογραμμίζω την ε, άριστη συνεργασία και την ισχυρή στήριξη που δώσατε σε σημαντικές προτεραιότητες του προπολογισμού. Νομίζω ότι εκφράζομαι και από πλευράς του κυρίου Έτιγκα, υπογραμμίζοντας ότι ήταν υποδειγματική η συνεργασία μας και προσβλέπουμε με βάση αυτή την θαυμάσια συνεργασία να καταλήξουμε επιτυχώς στην διαδικασία αυτή. Ω νέος Γενικός Διευθυντής για τον Προπολογισμό έμαθα πολλά τις τελευταίε εβδομάδε. Και ναι, μεν σημειώσαμε πολύ καλή πρόοδο. Επί της ουσίας δεν περίμενα εξάντε ότι θα συζητούσαμε για ταπεινώσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, αλαζονία, τέτοιους ε, συναισθηματικά φορτισμένους ε, όρους που αν εξετάσουμε την ουσία είναι ιδιαίτερα έντονη, αλλά ίσως όχι τόσο χρήσιμη. Ας δούμε σε ποιο σημείο ε, διακόψαμε τη συζήτηση μας ε, την προηγούμενη Δευτέρα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι εσείς και εμείς, Κοινοβούλιο και Επιτροπή, εργαστήκαμε για μια κατάσταση στην οποία σας αξίζουν συγχαρητήρια. Θα θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο ξεκίνησε προτείνοντας μια περικοπή 1,5 δι. Αλλά πολύ επιτυχώς ε, την απορρίψατε εντελώ αυτή την πρόταση και τώρα δεν συζητάμε περικοπέ, αλλά αυξήσει. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό επίτευγμα. Σημαντικότατο ο προπολογισμό για τον οποίο ε, έχετε πιέσει ούτως ώστε να είμαστε σε μια κατάσταση προκαταρκτικής συμφωνίας προκαταρκτική συμφωνία είναι ένα προβληματισμό που ανταποκρίνεται στι προσδοκίε και των ατόμων και τη οικονομία. Και νομίζω ότι κάνετε θαυμάσια δουλειά πιέζοντα για να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο και η Επιτροπή συνολικά σα είναι ευγνώμων στον ορίζοντα 2020 για παράδειγμα. Θα περάσουμε από έναν προπολογισμό 11,2 δι σε έναν προπολογισμό 12,3 δι. Αυτό είναι 1,1% περαιτέρω επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα, την ε, γνώση και την έρευνα, χάρη στην εργασία του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή σα Για τον έρασμο. Έχουμε μια αύξηση δαπανών από 2,3 δι σε νομίζω ότι σχεδόν είχατε συμφωνήσει διαπραγματεύσει σε περίπου 2,7 και εδώ χαρτίρια. Αυτό είναι αύξηση 400 εκατομμυρίων 400 εκατομμύρια, για να καταλάβετε τι σημαίνει, είναι 200.000 200.000 φοιτητές επιπλέον που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα έρασμο. Θα το θεωρούσα αυτό τεράστια επιτυχία. Επίσης, ήσασταν σε ένα σημείο όπου η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα ελάμβανε την πλήρη αύξηση που είχατε ζητήσει 116 εκατομμυρίων. Και αυτά ήταν νέα χρήματα, δεν ήταν απλώς προκαταρκτική χρήση πόρων. Και για τι προτεραιότητε, το μέσο γειτονία θα ελάμβανε μία αύξηση των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων, περίπου 100 εκατομμυρίων. Και η οικονομική βοήθεια στην Παλαιστίνη, την Ούνρα, Κύριε Γενική Διευθυντή, ο Πρόεδρος, οι διερμηνείς θα φύγουν πολύ σύντομα. Καλό είναι να επιθυμίζετε τι επετεύχθη, αλλά σε σχέση με αυτά που αναμένουμε, σε σχέση με αυτά που ακούσατε σήμερα το πρωί, εκεί θα θέλαμε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε, δεν το πετύχατε αυτό ακόμη. Αυτό ήταν στο σημείο ακριβώ που είπατε ότι δεν ε, πέτυχαν διαπραγματεύσει. Για να καταλαβαίνουμε, να σημειώσουμε, να καταλαβαίνόμαστε, να σημειώσουμε ότι χάρη στην θαυμάσια εργασία σα και την καλή συνεργασία έχουμε δυνατότητα να ε, επιτύχουμε 800 εκατομμύρια για τι προτεραιότητέ σα πάνω από αυτά τα οποία είχε προτείνει η Κομισιόν. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Είναι ουσιώδη πρόοδο ε, και θα πρέπει να είστε περήφανοι γι' αυτό. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το 15-3. Να σα υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή δεν είχε προτείνει το 15.3, ούτε το Κοινοβούλιο. Είναι κάτι που η Επιτροπή το ε, έβαλε στην πραγματεύση σε ένα σχέδιο συμβασμού. Είναι κάτι που ο δημοσιονομικός κανονισμός ε, το προτείνει ως κάτι καινούργιο. Είναι μια δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν αποδεσμευθείς πιστώσεις. Ε, όταν ακούω τι λέτε, είναι σαν να λέτε ότι απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός να γίνεται αυτό. Όχι, είναι μια δυνατότητα. Φυσικά ε, συμφωνούμε ότι είναι ιδιαίτερα λογικό, αλλά δεν είναι, υπάρχει κανένα αυτοματισμό. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο δημοσιονομικό κανονισμό. Και νομίζω ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει, γιατί όντω έχει έννοια. Το Συμβούλιο λέει ότι αυτή η ιδέα υπευλήθη τελευταία στιγμή, ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αξιολογηθεί. Εμεί από την πλευρά μα εκφράζουμε την απογοήτευσή μα για το πόσο ε, βράδυ μπορεί το Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο. Αλλά αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου. Η θέση τη Επιτροπή είναι ότι το μέσο αυτό είναι πολύτιμο και ότι όντω, όπω λέτε, θα ήταν πολύ καλό να το χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα συστηματικά. Θα πρέπει να το επιδιώξουμε λοιπόν όλοι αυτό. Αλλά επίση η Κομισιόν είπε ότι όταν θα γίνει αυτό και πώ θα γίνει και πώ θα ε, σημειωθεί είναι θέμα διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο σκελών τη αρχή του προπολογισμού. Καλωσορίζουμε τη θέση σα γι' αυτό, αλλά είμαστε ρεαλιστικοί, θέλουμε να επιτύχουμε καλό αποτέλεσμα. Επ' αυτού λοιπόν δεν μπορώ να δεσμεύσω σήμερα την ε, Επιτροπή. Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα για ένα προπολογισμό 165 δι σημειώσονται μεγάλη πρόοδο, δεν θα πρέπει να το ξανάτε. Πιέσα το Συμβούλιο να απομακρυνθεί από θέσει που εμεί ε, ω ε, Επιτροπή θεωρούσαμε πω ήταν ιδιαίτερα ατυχή, Αυτό είναι θαυμάσιο και η διαφορά που έχει μείνει μεταξύ των θέσεών σα δεν είναι διαφορά σε επίπεδο αρχή, γιατί είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία επί τη αρχή για τη χρήση του 15.3. Είναι διαδικαστική διαφορά. Και αφορά 200 εκατομμύρια σε έναν προπολογισμό 165 δις. Είναι σημαντικό ε, να το καταλάβει και το εκλογικό σώμα αυτό. Ότι τα πήγατε πολύ καλά, επιτύχατε πολλά και ότι τώρα αγγίζουμε σχεδόν κάτι οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Πραγματικά πολύ μικρές. Δεν θέλω να πολύ, πολύ περισσότερα για το δεχόμενο να αποτύχουν οι διαπραγματεύσει. Τότε θα περάσουμε στα προσωρινά 12 τιμόρια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα προπολογισμό που θα είναι παρόμοιο με τον προπολογισμό του 2018, με όλα τα μειονεκτήματα που ανέφερε ο πρόεδρο σε αυτή την κατάσταση, αλλά και με όλα τα μειονεκτήματα τη μη επίτευξη των καλών αποτελεσμάτων που προανέφερα. Θα ήταν κακό αποτέλεσμα κάτι τέτοιο. Αν η Ένωση δεν έχει προπολογισμό, τελευταία φορά που έγινε, όπω ξέρετε, ήταν το 1996. 1986, συγγνώμη, πριν από 32 χρόνια. Θέλετε να καταλήξουμε μια τέτοια κατάσταση. Ένα τόσο καλό προπολογισμό, ένα τόσο καλό προπολογισμό να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει προτεραιότητέ τη. Πρόεδρο, το σύστημα των 12 τιμωρίων λειτουργεί όσο δεν υπάρχει νέο προπολογισμό. Μα λέτε ότι θέλει χρόνο το Συμβούλιο για να εξοικειωθεί με το 15-3. Ίσως να του αρκέσει ο Ιανουάριο έτσι να εξοικειωθεί, να το συνηθίσει. Εμεί θεωρούσαμε ότι τρει μέρε ήταν ίσω λίγε, αλλά, αλλά τώρα έχουμε δύο εβδομάδε μέχρι να ψηφίσει ενδεχομένω το Κοινοβούλιο. Ίσως αυτό να επιτρέπει στο Συμβούλιο να μάθει καλύτερα το πώ λειτουργεί το 15-3 ούτω ώστε οι αρχές του προπολογισμού να ε, ε, συμφωνούν σε αυτά που λένε με τις διακηρύξεις των ε, αρχηγών κρατών κυβερνήσεων. Συμφωνούμε. Ε, φυσικά και μπορεί να βρεθεί λύση ε, στη διάρκεια του έτους. Ε, φυσικά, ε, έως ότου βρεθεί μια τέτοια λύση, οι δαπάνες θα είναι χαμηλότερες από τις αναγκές. Αν αυτό το επιθυμείτε, πρέπει να το σταθμίσετε εσείς ε, τα δύο θεσμικά όργανα στην ε, συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Να κάνω όμως ένα σχόλιο πρωτού κλείσω. Είμαι ευγνώμων για την εξαιρετικά μεγάλη υποστήριξή σας προς το άρθρο 15.3 και την ανάγκη να εφαρμοστεί. Θέλω όμως να υπενθυμίσω σε όλους ότι ούτε η Κομισιόν, ούτε το Κοινοβούλιο ήταν εκείνα τα θεσμικά όργανα που πρότειναν ε, αυτό το άρθρο στις ε, συνεισφορές τους. Και αυτό προσωπικά πρέπει να πω ότι με εκπλήσει λίγο. Κάτι το οποίο ε, η Κομισιόν το πρότεινε ως ε, λύση συμβιβαστική, ξαφνικά έχει γίνει το Άγιο Δισκοπότηρο. Και που θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι είναι τόσο σημαντικό που ακόμη και αν σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική, ε, εξετάζετε το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε από τις συνομιλίες το Δεκέμβριο. Αυτό είναι μια παρατήρηση ε, από τη δική μου πλευρά. Εντάξει, κατά τα άλλα βεβαίως επαναλαμβάνω ότι σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας και νομίζω ότι με τη σοφία που χαρακτηρίζει όλες τις πλευρές θα ε, καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία τον Δεκέμβριο. Που να σας πω την αλήθεια, ε, κοιτάζοντας το που βρισκόμαστε, ε, είναι μια συμφωνία για την οποία το Κοινοβούλιο μπορεί πραγματικά να είναι περήφανο. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είμαστε συμβολογραφικό γραφείο εδώ να μεταγράφουμε τις αποφάσεις που έχουν λάβει στο Συμβούλιο. Εμείς είμαστε πολιτικό θεσμικό όργανο και πρέπει να λογοδοτούμε και στους πολίτες. Λοιπόν, ο κύριο Γενικό ε, Εισηγητή, πολύ σύντομα. Και εγώ ευχαριστώ τους διερμηνείς για την υπομονή τους μιλητής, και για την υποστήριξή τους. Κύριε Κόπμαν, δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλει να εργαστεί το Κοινοβούλιο για να φτάσει στα προσωρινά 12 τιμόρια. Εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, κάνουμε τα πάντα και θα κάνουμε τα πάντα για να κλείσουμε ένα προπολογισμό που να είναι αξιοπρεπής. Η πρόθεση αυτής της Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και του Κοινοβουλίου και του Γενικού Εισηγητή δεν είναι να φτάσουμε στα 12 τιμόρια. Καμία τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να λέτε κάτι τέτοιο, ούτε μπορείτε να λέτε ότι μπροστά σε μια τέτοια προσφορά το κινδυνεύει το Κοινοβούλιο να οδηγήσει στην Ένωση στα 12 τιμωρία, γιατί δεν ισχύει αυτή η προσφορά που υπάρχει και να εξηγήσω γιατί επιμένουμε τόσο στο θέμα του άρθρου 15 παράγραφος 3, κύριε Γενική Διευθυντά. Καταρχήν, γιατί το άρθρο αυτό το ψηφίσαμε από κοινού και εμείς και το Συμβούλιο και γιατί είναι ένα διαθέσιμο μέσο και έγινε σημείο φετηρίως γιατί το Μάιο δεν είχαμε αυτό το εργαλείο. Ε, από τον Ιούλιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εφόσον το έχουμε θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και κλείνω για αυτά τα δύο στοιχεία το Συμβούλιο θέλει εμείς να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά. Θέλει να αναγκάσει το Κοινοβουλίο να κάνει αυτό που δεν είναι ικανό να κάνει ούτε τα κράτη-μέλη. Δηλαδή να χρηματοδοτήσει το μηχανισμό για την Τουρκία είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ε, να βάλει χρήματα για την έρευνα ε, και την ανάπτυξη. Προτιμούν να βάλουν νέο χρήμα και να παρουσιάσουν εμάς σαν αυτούς που ζητάνε χρήματα στα κράτη-μέλη. Και βλέπω τι λέει πω ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά περισσότερα κονδύλια από τα κράτη-μέλη, θέλουν περισσότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη. Είναι αυτοί που ξοδεύουν. Όχι, εμεί θέλουμε χρήματα που είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω δεν θέλω από τα κράτη-μέλη. Θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω εφιστάμενου πόρου. Γι' αυτό εμεί επιμένουμε τόσο για αυτού τους λόγου και το είπαν οι συνάδελφοι και το περιλαμβάνω και εγώ στην πρόταση που θα έρθει από την Κομισιόν η πρόταση αυτή θα πρέπει να ξεκινά από το ε, δεύτερα κοινά συμπεράσματα το σχέδιο, κοινό σχέδιο συμπερασμάτων και πρέπει να περιλαμβάνεται το 15.3 μια ερώτηση σε σχέση με τα 12 τιμόρια αν ε, επιτρέπετε, τι ε, δίνετε ε, στο μηχανισμό για την Τουρκία. Ποια είναι τα σχετικά κονδύλια. Απλώς ε, θα έχουμε το ποσό του 2018 αν δεν υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή θα πρέπει να δείξει κατανόηση το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Έχει λάβει μια θέση το Κοινοβούλιο και δεν αφιβάλλουμε ότι η Κομισιόν ε, θα βρει και τους κατάλληλους όρους, όμως ε, μέσω ε, των μέσων κοινωνικών δικτύσεων και με τους δημοσιογράφους που θα έρθετε σε επαφή, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε και να κάνετε και τις απαραίτητες επαφές με τις κυβερνήσεις σας για να ρωτήσετε αν υπάρχει επάρκεια μεταξύ των, του προϋπολογισμού και των δράσεων που προβλέπονται για την έρευνα. Στις 2.30 λέω πρόεδρε, πρόεδρος θα ξεκινήσουμε. 15h. Με συγχωρείτε. Λέει 2.30 το δικό μου το έγγραφο. On recommence à quelle heure On recommence à quelle heure À quelle heure À 15h. Alors, reprise des travaux. Θα ξεκινήσουμε εκ νέου τις εργασίες μας στις 3. Διακόπτεται η συνεδρίαση πρωινή.